Otwieram posiedzenie. Protokół wczorajszego posiedzenia. Ε, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως και άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα, ε, οπότε θέλω να ακούσω αν έχετε παρατηρήσεις επ' αυτού. Δεν ακούω κάτι τέτοιο, οπότε ε, υιοθετούνται τα πρακτικά. Ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ βασικό θέμα της σημερινής μας συνεδριάσεως. Είναι η ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.